και της Κίνας και καθεστώς οικονομίας της αγοράς. Πρώτος ομιλητής, ο κύριος Περντ Κλάνκε, συντάκτης της προφορικής ερώτησης. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, αναμφίβολα είναι πολύ σημαντικό εμπορικός εταίρος η Κίνα και για πολλές θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεράστια σημασία αυτό το εμπόριο. Το ζήτημα λοιπόν και το ερώτημα που συζητούμε έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όπως γνωρίζετε η Κίνα, και είναι πρόοδος αυτό, το 2001 προχώρησε με ένα πρωτόκολλο στην προσχώρηση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Στο άρθρο 15 του σχετικού πρωτοκόλλου προσχώρησης έχει προβλέψει μια 15 ετή περίοδο μετάβασης με σταδιακή κατάργηση, κατάργηση των μέτρων dumping και επιδοτήσεων. Εκπνέει λοιπόν αυτή η περίοδος της προσαρμογής και πρέπει να αναλογιστούμε τα περαιτέρω. Διότι είναι αμφιβολό ότι η διαδικασίες για την αντιμετώπιση του ντάμπινγκ και των επιδοτήσεων είναι σχετικές με τη στάση και τη συμπεριφορά της Κίνας. Κατά 80% είναι διαδικασίες ε, που απευθύνονται στην Κίνα αυτές οι διαδικασίες και κατά των επιδοτήσεων γιατί στρεβλώνουν τις τιμές και αφορούν τον σχηματισμό τιμών από τρίτε χώρες αυτές τι δικασίες. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε στις 11 Δεκεμβρίου με την εκπνοή αυτή τη μεταβατική περίοδου τι συνέπειε έρχονται. Και αν αναγνωρίσετε το καθεστώ οικονομία τη αγορά για την Κίνα ή αν πρέπει να αναγνωρίσετε. Ταυτόχρονα έχουμε ένα μοχλό προστασίας ε, για τα δικά μας προϊόντα που δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε ε, χωρίς συζήτηση. Πιστεύω ότι θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να μελετήσουμε τα θέματα αυτά, το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο μαζί με το Κοινοβούλιο τόσο άλλως θα πρέπει να ε, συνεννοηθούν. Και γι' αυτό διαρωτώ με και πώς έφυγαν από τα χέρια μας αυτά τα 15 χρόνια, γιατί δεν δουλέψαμε νωρίτερα να προετοιμαστούμε. Τρεις είναι οι επιλογές. Ή να αφήσουμε να προχωρήσει αυτοματοποιημένα αυτή η διαδικασία ώστε να αναδοθεί το καθεστώς οικονομίας της αγοράς στην Κίνα και έτσι να σταματήσουν αυτομάτως ε, οι δυνατότητες, δηλαδή να παραιτηθούμε ουσιαστικά από τη δυνατότητα επιβολής μέτρων κατά του ντάμπινγκ και κατά των ε, επιδοτήσεων, πράγμα το οποίο έχει ήδη πράξει η Αυστραλία με κακέ συνέπειε, γιατί δεν έχει, δεν έχει στα χέρια τη αυτό το μέσον ε, αντίδρασης. Δεύτερη επιλογή, ένα περιφραστό όχι, άρα αμέσως προξενείται προσφυγή στον ΠΟΕ και τρίτον, και αυτό είναι η δυνατότητα που προσφέρει και το πρωτόκολλο, με ένα περιθώριο ε, χειρισμών που επιτρέπει γιατί προβλέπει εναλλακτικέ μεθόδους σε σχέση με την ε, διαμόρφωση τιμών από τρίτα κράτη όπου ε, καλούνται εκείνα τα κράτη να έχουν την υποχρέωση απόδειξη ότι δεν προβαίνουν σε ντάμπινγκ ή σε παράνομες επιδοτήσεις. Άρα μπορούμε και μετά τις 11 Δεκεμβρίου, εάν επιλέξουμε αυτή την τρίτη λύση, να έχουμε έναν ικανοποιητικό μηχανισμό προστασίας. Φυσικά αυτό σημαίνει ότι θα προβούμε σε συνομιλίε με τους Κινέζους εταίρους για να καταλήξουμε σε μια λογική λύση. Συνομιλίε που τόσο ή άλλω θα πρέπει να αναπτύξουμε γιατί δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε την υπερπαραγωγή μέσω των κρατικών επιδοτήσεων παροιόντων τα οποία στη συνέχεια θα ε, κατακλείσουν τις ευρωπαϊκές αγορές όπως συμβαίνει τώρα σε έναν βαθμό. Υπάρχει μεγάλη άλλωστε διαδήλωση ε, που έχει προβλεφθεί όπως ξέρετε για τον τομέα του Χάλιβα για τον Φεβρουάριο στις Βρυξέλλες γιατί ο κόσμος αντιδράει όπως ξέρετε. Ή πρόκειται για επιδοτήσεις στον τομέα του χάλιβα από τις οποίες δεκυβεύονται θέσεις εργασίας. Πρέπει λοιπόν πολύ προσεκτικά να αναλύσουμε τι συνέπειες των τριών επιλογών που σας περιέγραψα και να κάνουμε την επιλογή ώστε να μην κινδυνέψουν και θέσεις εργασίας αλλά και να ενισχυθεί η βιομηχανική ανάπτυξη στην Ευρώπη 20% του ΑΕΠ που πρέπει όχι μόνο να διατηρηθεί αλλά και να ενισχυθεί, πάντως όχι να αποδυναμωθεί. Ε, από τον Απρίλιο του 2014 το Συμβούλιο δεν μεταρρυθμίζει τα μέσα προστασίας και από την άλλη βλέπουμε να προωθεί το ζήτημα της αναγνώρισης του καθεστώτος της οικονομίας αγοράς στην Κίνα. Δεν είναι σαφή η θέση του λοιπόν. Απαιτείται να τοποθετηθεί ξεκάθαρα και γι' αυτό ζητώ και από εσά, κυρία Επίτροπε να μας πείτε τι θέλετε. Πότε θέλετε να καταθέσετε προτάσεις και τι περιεχόμενο θα έχουν αυτές οι προτάσεις. Ähm, Ο ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον κύριο Λάγκε που μου δίνει τη δυνατότητα να συζητηθεί αυτό το θέμα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με όλους. Για να σας ενημερώσω και όλους που βρισκόμαστε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να διευκρινίσω ότι το ερώτημα δεν είναι κατά πόσον η Κίνα είναι μια ε, χώρα όπου υπάρχει η οικονομία της αγοράς ή όχι. Όχι. Το ερώτημα είναι κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζει το ντάμπινγκ, εάν υπάρχει dumping, σε έρευνε ε, καταπολέμησης του dumping. Και ο λόγο είναι ακριβώ αυτή η εκπνοή τη 15ετού περίοδου που είχε προβλεφθεί στο πρωτόκολλο ε, προσχώρηση τη Κίνα στον ΠΟΕ, όπω ε, περιέγραψε ο κ. Λάγκε, κάτι το οποίο θα έχει επιπτώσεις για τη βιομηχανία μας. Το 38% των εισαγωγών μας από την Κίνα επηρεάζονται, αλλά αυτό έχει τεράστια σημασία για ορισμένες επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξελογεί τι διάφορε επιλογέ που έχει στη διάθεσή τη. Πρώτα απ' όλα, μία δυνατότητα είναι να μην αλλάξουμε την νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην αλλάξει ε, λοιπόν ο τρόπο υπολογισμού του dumping στι 11 Δεκεμβρίου του 2016. Το οποίο όμως θα έχει επιπτώσεις και πιθανώς να προσβληθεί και νομικά. Αυτό θα έχει κόστος επίσης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε θέσεις εργασίας. Το κόστος είναι σχεδόν αδύνατον να το υπολογίσουμε εκ των προτέρων. Υπάρχει επίση ο κίνδυνο να θεωρηθεί ότι σε αυτήν την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παραβιάσει τι υποχρεώσει τη στο πλαίσιο του ΠΟΕ με πιθανεί οικονομικέ επιπτώσει. Υπάρχει μια νομική άποψη που λέει ότι, το ότι κάποιες από τις προβλέψεις του πρωτοκόλλου δεν θα ε, εκπνεύσουν, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του σίγουρα θα εκπνεύσει. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε τη συνέχιση της διεθνής πολιτικής, αλλά αυτό θα είχε δυσμενείς επιπτώσει για κράτη-μέλη και για ευρωπαϊκέ επιχειρήσει. Μια τρίτη επιλογή θα ήταν να θεωρηθεί η Κίνα ως καθεστώς οικονομίας της αγοράς, ταυτόχρονα όμως θεσπίζοντας μέτρα για να αντισταθμίσουμε τις πολλές ε, ε, ε, καταστάσεις που υπάρχουν στην κινέζικη οικονομία, στρεβλώσεις που υπάρχουν στην κινέζικη οικονομία. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε προσεκτικά τις επιλογές μας, όποια και να επιλέξουμε τελικά, Σα διαβεβαιώνουμε ότι θα υπάρχει ένα ισχυρό εργαλείο για το αντι-dumping, το οποίο θα προστατεύει τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει ταυτόχρονα ε, σε συμφωνία με τι διεθνεί μα υποχρεώσει. Πρέπει να αλλάξει η μεθοδολογία ε, του υπολογισμού του αντι-dumping όταν λήξει το Δεκέμβριο η περίοδο του πρωτοκόλου, αλλά αυτή η δυνατότητα αναλογικού, ε, αναλογικού υπολογισμού που είχαμε μέχρι στιγμής δεν θα μπορέσει να συνεχιστεί. Τα θέματα αυτά είναι πολύ τεχνικά, είναι δύσκολα, αλλά έχουν σημαντικέ επιπτώσει. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει μια αξιολόγηση αντικτύπου. Ε, Ει βάθο, αυτό που έχετε λάβει ω αξιολόγηση αντικτύπου είναι απλώ το προσχέδιο. Θα ενημερώνουμε τακτικά την Επιτροπή του Κοινοβουλίου την Αρμόδια, γιατί επιθυμούμε μια συνεργασία με διαφάνεια μαζί σας. Τώρα όσον αφορά την συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, και εδώ είναι σημαντικό το θέμα, έχουμε ήδη ξεκινήσει επαφές με τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μας έχουν εκφράσει τις απόψεις τους. Αρχικά φαίνεται κάναμε άλλο μία μελέτη για τον αντίκτυπο που θα είχε στις ε, ε, θέσεις εργασίας και διαπιστώνουμε ότι πιθανώς, εάν αλλάξει λοιπόν ο τρόπος υπολογισμού, ε, σε, στο συνηθισμέ, και πάμε προς το συνηθισμένο τρόπο υπολογισμού του αντι-dumping, και έχουμε επίσης υπολογίσει ότι δεν θα συμβεί στο σενάριο που δεν θα λάβουμε μέτρα αντισταθμιστικά. χειρότερο σενάριο περιμένουμε 34.000 έως 74.000 εργασία θα χαθούν. Η μελέτη επίσης μας λέει ότι μακροπρόθεσμα αυτοί οι αριθμοί μπορεί να ανέλθουν από 73 μέχρι 88.000. Δεν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας βέβαια και τις επιπτώσεις που θα είχε σε άλλους κλάδους της οικονομίας που συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις τις οποίες αφορά το προηγούμενο αριθμό και τότε μιλάμε για 63.000 έως 210.000. Αυτή η αριθμή είναι μεγάλη, αλλά μικρότερη από ε, μελέτες άλλων οργανισμών όπως το ε, Policy Institute στην Ουάσιγκτον. Ε, και βέβαια υπάρχει δυνατότητα λήψης αντισταθμιστικών μέτρων, αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε τη, συμφωνία, τη σημασία αυτών των κινδύνων. Έχει τεθεί επίσης το ζήτημα του συντονισμού με άλλες χώρε. Και πράγματι έχουμε ξεκινήσει επαφέ αλλά βέβαια είναι γνωστό ότι οι νομικές υποχρεώσεις των κρατών μελών του ΠΟΕ πρέπει να γίνουν σεβαστές. Κάποια κράτη δεν χρειάζεται, κάποιες τρίτες χώρες δεν χρειάζεται να τροποποιήσουν την νομοθεσία τους. Κάποιες χώρες μπορούν να αλλάξουν τις αποφάσεις τους και την πολιτική τους σε πέντε λεπτά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί η τροποποίηση της νομοθεσίας. Αυτό είναι κάτι που μας ε, κάνει ε, να βρισκόμαστε σε μια ξεχωριστή ε, θέση και όχι για παράδειγμα όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε. Γιατί κάποιες χώρες δεν είχαν ήδη αναγνωρίσει το καθεστώς του, της, αγοράς, της οικονομίας της αγοράς στην Κίνα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα, αλλά θα χρειαστεί αλλαγή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, όπου βεβαίως θα ακολουθηθεί η διαδικασία η συνήθις και το, η πρόταση θα έρθει από την Επιτροπή προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα συνομοθετήσουμε. Βεβαίω η συζήτηση ως τότε θα συνεχιστεί και ευχαρίστω να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ο κύριος Βίγκλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί ε, συνάδελφοι, αγαπητοί επίτροπε. Το θέμα των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Κίνας ε, δεν θα πρέπει να μας σταματήσει από το να λέμε ότι δεν πληρεί ακόμη τα κριτήρια για το καθεστώς της οικονομικής αγοράς. Έχουμε την νομική πτυχή που πρέπει να λάβουμε υπόψη, ο αυτοματισμός, η αυτοματοποίηση για την τροποποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ε, δεν είναι αυτόματη η διαδικασία χωρίς καθεστώτος ε, της ε, οικονομικής αγοράς. Επίσης υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Θέλουμε από την Κομισιόν μελέτη αντικτύπου πλήρη, διεξοδική. Έχουμε και το γεωπολιτικό πλαίσιο στο αφορά τη στρατηγική εταιρική σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνα. Χρειάζεται περισσότερη συνεργασία, λιγότερο ανταγωνισμό. Επίση, Θέλουμε συμβατές ε, και προς τον ΠΟΕ και νομικά ε, ε, σωστές λύσεις. Και σε ό,τι αφορά το μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Το σύστημα θα πρέπει να κρίνει και τις διαφορές με την Κίνα στο μέλλον. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και η επιχειρηματική κοινότητα τη Ένωση θα πρέπει να συμμετέχει. Θέλουμε ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα, ώστε οι δυνάμει αγορά να ορίζουν τον ανταγωνισμό και να μην έχουμε κρατικέ παρεμβάσει. Ευχαριστώ. Thank you very much. ευχαριστώ. 15 χρόνια τώρα ξέραμε ότι το καθεστώς της οικονομίας ε, της αγοράς θα έπρεπε να εγκριθεί για φέτος για την Κίνα, αλλά η Επιτροπή δεν προχώρησε καμία απόφαση και δεν έχει καμία σαφή στρατηγική σχεδιάση. Ούτε κι εμείς βέβαια ξυπνήσαμε την ε, Επιτροπή από το λιθαργό τη. Τώρα ελπίζω ότι θα ξεκινήσει ένα σοφρό διάλογο με το Κοινοβούλιο, τα κράτη-μέλη, ε, το βιομηχανικό κλάδο, του εργαζομένου και βέβαια την Κίνα. Γιατί θέλουμε καλέ σχέσει με την Κίνα. Ξέρουμε ότι η Κίνα θεωρεί πως θα πρέπει αυτομάτως να τη χωρίζεται το καθεστώς ε, της οικονομίας αγοράς το Δεκέμβριο. Ταυτόχρονα όμως φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεται εκείνα ότι και εμείς έχουμε σαφείς προσδοκίες το 2001 είχαμε σαφείς προσδοκίες ότι ως το, 26, ως το, 16 θα είναι πραγματική οικονομία αγοράς η Κίνα. Και από αυτά που μας λέει η Επιτροπή δεν είναι πραγματική οικονομία της αγοράς, επομένως δεν μπορεί να της χορηγηθεί αυτομάτως το καθεστώς αυτό. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην Κίνα την υπερπαραγωγή της να την διοχετεύει σε ευρωπαϊκές ε, αγορές για να απαλλαγεί από αυτήν. Και όπως είπε υπάρχουν 52 διαφορετικές έρευνες για θέματα dumping, δεν είναι το μόνο πρόβλημα δηλαδή ο κλάδος του Χάλιβα. Πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι δεν είναι προστατευτισμός το να αμήνεται κανείς έναντι του αθέμητου ανταγωνισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται διακαώς ένα πιο σύγχρονο καθεστώς και μέσα προστασίας. Όρο εκ των όνων για την υποστήριξη τουλάχιστον για μένα, του καθεστώτος οικονομίας αγοράς για την Κίνα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ εκ μέρους του ECR. Για ένα λεπτό, κυρία Μακκλάρκιν. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το καθεστώ οικονομία αγορά για την Κίνα είναι ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα που θα έχει να αντιμετωπίσει φέτο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πολλέ πτυχέ που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κατά τη συζήτηση αυτή και πρώτα απ' όλα με βάση και τη γνωμοδότηση νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γνωρίζει ποιες είναι δεσμεύσεις της δυνάμει του δικαίου του Διεθνούς Εμπορίου του ΠΟΕ με το πρωτόκολλο 15α προσχώρησης της Κίνας στον ΠΟΕ. Ταυτόχρονα γνωρίζω και εγώ πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό δεδομένου ότι και στη δική μου τη χώρα η Χαλιβουργία έχει γονατίσει και μπορεί ποτέ να μην ανακάμψει και πολλά ζητήματα θα πρέπει να επιληθούν σε συνθήκες ε, θεμητού ανταγωνισμού. Οτιδήποτε λοιπόν και να προτείνει το πρωτόκολλο, το ε, δίκαιο αντινάπινγκ της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας επιτρέπει και θα πρέπει να μας επιτρέπει την δυνατότητα ακόμη να αντιμετωπίσουμε αθέμητες ε, πρακτικές και παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μιλήσει λεπτομερώς για τις συνέπειες από την αλλαγή της μεθοδολογίας σε σχέση με τους δασμούς αντινάπινγκ αλλά και τα μέσα που έχουμε για άμυνα έναντι των αθέμητων πρακτικών. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους των φιλελευθέρων, η κυρία Σχάκη. Δύο λεπτά. Πρόεδρε, συνάδελφοι, ε, κύριε Επίτροπε, το dumping προϊόντων στην αγορά μας με τιμές κάτω του κόστους δεν πρέπει να επιτρέπεται και πρέπει να αντιμετωπιστεί με αντίμετρα. Πώς όμως θα εξασφαλιστεί αυτό όταν εκπνέει το σχετικό πρωτόκολλο με τη μεταβατική διάταξη που είχε υπογραφεί πριν από 15 χρόνια για την προσχώρηση της Κίνας στην ΠΟΕ το θέμα δεν είναι να πιστεύουμε εμεί ότι η Κίνα έχει οικονομία τη αγορά ή ότι τηρεί του όρου τη τη προσφορά και τη ζήτηση, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει βέβαια, αλλά πώ θα αντιμετωπίσουμε τι αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ ενό πολύ σημαντικού εμπορικού εταίρου. Η ομάδα μου πιστεύει ότι θα πρέπει το περίπλοκο αλλά και τεχνικό αυτό θέμα να το αντιμετωπίσουμε με μεγάλη ψυχραιμία. Κάποιοι ήδη τοποθετούνται συγκινησιακά ή προσπαθούν να αξιοποιήσουν την ε, ευκαιρία αυτή για να μιλήσουν για προστατευτικά μέτρα. Ε, αλλά μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη έχει και εξαγωγές όπως και εισαγωγές. Και άρα δεν πρέπει να κοιτούμε μόνο τα εισερχόμενα προϊόντα. Νομίζω ότι χρειάζεται μια δεξιοδική αξιολόγηση συνεπειών και της πρόσβασης αγοράς και ένα σύστημα εμπορίου, ιδιαίτερα σχέση με την Κίνα, έχει κέρια σημασία και εμείς να κοιτάξουμε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης να τηρούμε τα όσα κηρύττουμε και να είναι πάντοτε σύμφωνες με τις διατάξεις του ΠΟΕ οι ε, ρήτρε μα και οι κυρώσει μα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε αμυντικά μέσα για τι επιδοτήσει ή το τάμπιν ή οτιδήποτε άλλη, α θέμα είναι ότι ή το dumping ή οποιαδήποτε άλλη αθέμητη πρακτική μπορεί να υιοθετεί η Κίνα ή άλλος εταίρος σε τελευταία ανάλυση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υιοθετει η κινα η αλλο εταιρος σε τελευταια αναλυση πιστευω οτι ε, θα πρέπει να δρούμε έγκαιρα και αποφασιστικά και να μην αφήνουμε τελικά να αποφασίζει μόνο η διαδικασία διευθέτησης διαφορών του ΠΟΕ. Ευχαριστώ πολύ για ένα λεπτό εκ μέρους της αριστεράς ο κύριος Σόλτς. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση δεν θα πρέπει να εξαντληθεί στο αν είναι η οικονομία της αγοράς η κοινή παγκοσμιοποίηση, απαιτεί πολιτική ρύθμιση των αγορών. Είναι σημαντικό λοιπόν ε, να σημειώσουμε ότι έχει προχωρήσει 12% η αύξηση των μηνιαίων μισθών κατέτος στην Κίνα και πρώτα η Κίνα Βλέπουμε να έχει υψηλότερου μισθού ακόμη και από, πολύ, από γνωστά μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρουμανία, Τσεχία κτλ. Αυτό σημαίνει σημαντικέ συνέπειε για τι εισαγωγέ ε, από την Κίνα. Πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το τάμπινγκ, να διαφυλάσσουμε τι θέσει εργασία τόσο στην Ευρώπη αλλά και στην Κίνα. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να, κάνουμε, να ερχόμαστε αντιπαράθεση, αλλά να κοιτάξουμε να συνεργαστούμε με την Κίνα και γι' αυτό ερωτώ το εξή, κύριε Επίτροπε, με μια συγκεκριμένη πρόταση μπορούμε να προχωρήσουμε πέραν των όσων προτείνουν τα όρια του ΠΟΕ για να συνάψουμε μια διμερή συμφωνία αντι-dumping με την Κίνα και κανόνες οι οποίοι θα διαμορφώνουν υγιείς συνθήκες διαμόρφωσης των ε, τιμών ώστε να αποτρέπεται και το κοινωνικό dumping. Ευχαριστώ πολύ για δύο λεπτά εκ μέρους των προσήμων ο κύριος Μπιουτικόφερ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε και κύριοι. Η Κίνα δεν είναι η οικονομία της αγοράς, πλην όμως, λέει η κυβέρνησή τη θα πρέπει να μας αναγνωρίσετε ως οικονομία της αγοράς, διότι πρώτον η οικονομική ε, πραγματικότητα είναι αυτή ε, και διαφυσβήτητη και επίσης μας το έχετε υποσχεθεί. Ναι, τους το έχουμε υποσχεθεί, αλλά η Κίνα ετήρησε αυτά που είχε υποσχεθεί πριν από μία δέκα πενταετία. Τώρα δεν θέλω να κάνουμε συμψηφισμούς, αλλά είμαι διατεθειμένος μία μη οικονομία της αγοράς να την αναγνωρίσω ως οικονομία της αγοράς στο βαθμό που δεν βλάπτει τη δική μας οικονομία της αγοράς ε, σοβαρά και ε, με μεγάλες ζημιές ε, λόγω της συμπεριφοράς. Υπάρχει τέτοια απειλή για τέτοιες ζημιές βεβαίως. μέχρι 3,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας ε, απειλούνται. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει μπορεί να είναι 200.000. Γιατί και 200.000 να είναι θα πρέπει να μας θορυβεί αυτό και είναι πάρα πολλέ. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσε θέσει διακυβεύονται. Γι' αυτό πρώτον θα πρέπει να κάνουμε μια πλήρη μελέτη αντικτύπου και συνεπειών. Βεβαίως θα ήθελα να προειδοποιήσω ούτε εσεί, κυρία Επίτροπε Ε, δεν ε, ε, έχετε ανισχύσει από το 1,38% των συναλλαγών που αφορά το dumping. Αλλά αυξάνονται τα πλεονάσματα στην Κίνα και πιέζουν την αγορά των εξαγωγών και δεν μπορούμε να δηλώνουμε ικανοποιημένοι με αυτό το ποσοστό. Θα πρέπει να προνοήσουμε. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θέλουμε να είμαστε αφελείς εις βάρος θέσεων εργασίας δεν θα πρέπει ανεφόρον να ανταποκριθούμε στα όσα ζητάει η Κίνα. Να κάνουμε προσφορά, να τις δώσουμε καθεστώς οικονομία της αγοράς εάν ταυτόχρονα υπάρξουν και ε, αποτελεσματικά εργαλεία κατά του ντάμπινγκ. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Διαφορετικά στο Κοινοβούλιο δεν πρόκειται να βρείτε συνένεση. Ευχαριστώ κύριε Μπιουτικόφερ. Από την ομάδα του ο κύριος Μπορέλη για μισή λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Στις 11 Δεκεμβρίου φέτος η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εκφράσει μια σαφή θέση η οποία να είναι αποφασιστική σημασία σε σχέση με το καθεστώς οικονομίας της αγοράς για την Κίνα. Εάν λάβουμε υπόψη και, την, ε, και το επαγγελματικό τομέα και την απασχόληση θα πρέπει να δούμε ποια θα οριστεί ως θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι πιο διαφανής και αποτελεσματική αυτή η πρόκληση. Θα πρέπει να ζητήσουμε περισσότερο για το δικό μας επιχειρηματικό κόσμο. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ένα έγγραφο το οποίο απέχει από τις εκτιμήσεις που έκαναν οι ίδιες επιχειρήσεις για τη θέση σε κίνδυνο ε, θέσεων εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά το ζήτημα. Η Επιτροπή θα πρέπει να διαπραγματευτεί πολύ σοβαρά και να βάλει όλο το πολιτικό βάρος της Ευρώπης για να αποστείλουμε προς την Κίνα ένα σαφές μήνυμα. Δεν θα πρέπει να δεχτούμε τις απειλές προσφυγής των ΠΟΕ. Έτσι κι αλλιώς κάτι τέτοιο δεν αρμόζει ούτε στους Κινέζους. Για... Λεπτό, ψωνόματος τη ομάδα τη κυρία Κάπελ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Ε, ο φτηνός χάλιβας με υψηλές επιδοτήσεις από την Κίνα κατακλείζει την ευρωπαϊκή αγορά και ευθύνεται για την κρίση στη χαλιβουργία που έχει οδηγήσει σε μετεγκαταστάσεις και απώλεια ε, θέσεων εργασία κατά χιλιάδες. Από το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει 16 ε, προσφυγές επί 6 αφορούν την Κίνα για τη χαλιβουργία και έχει ε, βάλει ε, πρόστιμο και ε, δασμούς μέχρι 25% σε συγκεκριμένα προϊόντα ε, χάλιβα ψυχρής ελάσσεως. Παρ' όλα αυτά η Κίνα τώρα ε, έχει την αξίωση μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου να έχει αναγνωριστεί ως οικονομία της αγοράς από τον ΠΟΕ. Αυτό σημαίνει ότι για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα είναι πολύ πιο δύσκολο να επιμείνουν για να υπάρξει δίκαιη ε, μορφή ανταγωνισμού είναι υψηλό το κόστος ε, εργασίας και ενέργειας στην ε, Ευρώπη. 3,5 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης ή 2% του ΑΕΠ κινδυνεύουν και απειλούνται. Άρα χρειάζεται όλοι να δράσουμε από κοινού. Ο Πρόεδρος διακόπτει την κυρία Κάπελα, αλλά ένα λεπτό δεν μπορώ να σας αφήσω ε, παραπάνω από ένα λεπτό και 15 δεύτερα. Τώρα. Ως μία γεγραμμένος για ένα λεπτό ο κύριος Κορβεμίκε. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα συμβεί αν εμείς ε, ε, θεωρούμασταν ε, μία, μη οικονομία αγοράς. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι τιμές στον τομέα της ενέργειας είναι εντελώς τεχνητές, άρα δεν είμαστε οικονομία της αγοράς. Εάν το North Stream ισχύσει, τότε έχει καλός. Αλλά οι πολιτικοί αποφασίζουν και θα ήθελα να ρωτήσω τους ε, σοσιαλιστές που είναι υποκριτές και που παρίστανται στην αίθουσα να μην λαλάβουν υπόψη αλλά να μην λάβουν υπόψη μόνο το μεγάλο κεφάλαιο. Θα ήθελα να σας υποβάλω μία ερώτηση. Τι θα συμβεί εάν η Κίνα αποφασίσει του χρόνου ή φέτος το ε, ε, τα Χριστούγεννα ότι θα πρέπει να δώσει σε κάθε παιδί ένα δώρο 100 ευρώ. Αυτό τι θα προστατεύσει τα, τα παιδιά από το να πληγούν από διάφορες ασθένειες, για παράδειγμα. Κασπάρη. Εξαιρετικό κύριε Πρόεδρε, για τη δική μας πολιτική ομάδα, αυτό που είναι σημαντικό είναι και μετά τον Δεκέμβριο να προστατεύσουμε τους υπαλλήλους μας, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις μας από αυτά τα κινέζικα προϊόντα. Η Επιτροπή λοιπόν εδώ μας αναφέρει διάφορες εναλλακτικέ, τις οποίες ανέφερε εξάλλου η Επίτροπος, όσον αφορά τις πιθανές ε, επιπτώσεις, τι πρέπει να περιμένουμε. Έχουμε όμως ε, εμείς στην Ευρώπη ρυθμίσεις, ε, έχουμε νομοθεσία, έχουμε την οικονομία της αγοράς και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι οι Κινέζοι βεβαίως δεν είναι το σύστημά τους οικονομία της αγοράς, αλλά την άλλη ώρα έχουν ένα εντελώς ανεπαρκές και αναποτελεσματικό σύστημα. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, το αποτέλεσμα είναι ότι όλα αυτά τα προϊόντα πλήττουν την ευρωπαϊκή οικονομία. Και εμείς θα πρέπει να βρούμε τρόπους να προστατευτούμε. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το 2000 όταν ήταν έτοιμη να μπει στον ΠΟΕ η Κίνα, υπήρχε μια προφορική ερώτηση που απέφθηνε εκ μέρους της Επιτροπής Ήτρε προς την Επιτροπή. Ήταν ε, συνάδελφος Μάν τότε. Και επρόκειτο για την τήρηση των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει η Κίνα να τηρήσει αυτές τις υποχρεώσεις της ε, που είχε δεχθεί πριν προσχωρήσει στον ΠΟΕ. Ευχαριστώ πολύ. Η συνάλφος Μόσκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι είμαστε ικανοποιημένοι για αυτή τη συζήτηση γιατί οι Κινέζοι θα ετοιμαστούν για τη θέση μας. Δεν υπάρχει αυτοματισμός και μονομέρεια στην πρόσβαση στην οικονομία αγοράς. Οι πιέσεις των προηγούμενων μηνών οδήγησαν την ε, Κομισιόν να αναβάλει την απόφαση για το δεύτερο εξάμεινο του 2016. Ελπίζω να το χρησιμοποιήσουμε αυτό για να δούμε ποιοι θα είναι οι αντίκτυποι έτσι ώστε η Κίνα να ακολουθήσει τις κατευθυντήριες γραμμές και να βρει και εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Όμως θα πρέπει να λάβουμε μία απόφαση ζωτικής σημασίας τη στιγμή που είχαμε 15 χρόνια στη διάθεσή μας για να οικοδομήσουμε μία χρήσιμη στρατηγική. Άρα βιαζόμαστε, βιαζόμαστε ιδιαίτερα γιατί δεν υπάρχει τρόπος επιμερισμού των κινδύνων έτσι ώστε να μην Είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τη, τους δασμούς και το dumping που επιβάλλουν οι Κινέζοι. Δεν ε, πρόκειται για ιδεολογικούς περιορισμούς. Θα πρέπει όμως να υπάρχει πλήρης ισότητα των πάντων και από τα δύο συμβαλόμενα μέρη. Daniel Dalton. Εγώ προέρχομαι από τα West Midlands, όπου είχαμε, είχαμε πλεόνασμα την Κίνα Τρία δις στερλίνες. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν πραγματικά επιδοτήσεις. Ναι, το κράτος παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία, ναι, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την Κίνα όπως όλους τους άλλους. Αν είμαστε προστατευτικοί, τότε θα ανταπαντήσουν βία και αυτό θα έχει επιπτώσεις στις θέσεις εργασίας. Η Κίνα διάλεξε τον ΠΟΕ, έπαιξε με τους δικούς μας όρους. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να ανταποκριθούμε στις ε, υποχρεώσεις μας. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις παραμέτρους του ΠΟΕ για να αντιμετωπίσουμε το dumping από πλευράς Κίνας. Και μετά θα πρέπει να αναζητήσουμε μία ε, συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με την Κίνα. Θα πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στον ΠΟΕ και εμείς οι ίδιοι. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Σαρνές για ένα λεπτό δεν πρόκειται απλώς για ένα δύσκολο θέμα και λεπτό. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό για την έρευνα, για την οικονομία μας, για τη βιομηχανία και για τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Και δεν πρέπει να λαμβάνεται και κλεισμένο των θυρών. Χρειάζεται μια δημόσια ανοιχτή συζήτηση, καθότι πρόκειται για πολύ σημαντικά θέματα. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι αυτόματη η απάντησή μας. Η Κίνα πληρεί τα κριτήρια της οικονομίας αγοράς. Το ξέρουμε όλοι ότι η απάντηση είναι όχι. Όσο λοιπόν δεν περάσει από μεταρρυθμίσεις η Κίνα, όσο ο ανταγωνισμός δεν θα είναι θεμητός, όσο δεν θα παίζουμε επίσης όρεις με την Κίνα, θεωρώ ότι δεν πρέπει να τις δώσουμε το καθεστώς της οικονομίας αγοράς. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ για ένα λεπτό ο William Earl of Dartmouth. Ευχαριστώ πολύ. Η Κίνα βεβαίως ζητάει το καθεστώς της οικονομίας αγοράς. Είναι όμως ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ε, προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι οι εξαγωγές της Κίνας είναι πολύ περισσότερες από αυτές του Ηνωμένου Βασιλείου. Και χωρίς να είναι κράτος μέλος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας αφήσουμε το χάλιβα. Ξέρετε το dumping που γίνεται χάνονται θέσεις απασχόλησης και βεβαίως στο Ηνωμένο Βασίλειο βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουμε σοβαρές προκλήσεις. Και αυτό σε ισχύει για όλη τη βιομηχανία. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει την δυνατότητα να επιβαλλει σμούσαν την αντι-dumping στην Κίνα και βλέπετε ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά θα μπορούσε να είναι διαφορετική η κατάσταση στην περιοχή των West Midlands, παραδείγματο χάρη. Σύμφωνα με τις αρχές Ευρωπαϊκή Ένωσης, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, 3,5 εκατομμύρια θέσεων απασχόληση κινδυνεύουν να χαθούν. Βλέπω ότι υπάρχει μια μπλε κάρτα από τον David Martin. Τη δέχεστε? Πιστεύετε, ακούγοντας ε, το τι ανέφεραν ε, σήμερα η συντηρητική και τον χαιρετισμό του ε, Πρωθυπουργού έντατη της Κίνας, αν εμείς δεν ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα εφαρμόζαμε επιδοτήσεις αντι-dumping κατά της Κίνας, δασμούς, με συγχωρείτε. Κύριε Μάρτιν, σας εκτιμώ ιδιαίτερα αλλά εάν λέτε ότι ο Πρωθυπουργός ε, στην ουσία είναι αδύναμος και δεν προωθεί τα βρετανικά συμφέροντα και είναι μικρόψυχος έναντι των συμφερόντων μας και έναντι της Κίνας, τότε θα πρέπει να πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Σαφής η απάντηση. Ο Ζόλιο εξαφάζει για ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, γνωρίζετε το χάρτη της Αμπάνας. Δεν ξέρω. Υπεγράφει το 48 παρόλα αυτά μετά από πρωτοβουλία του ΟΙΕ, έτσι ώστε να καθοριστούν νέοι κανόνες για την ενδυνάμωση της ειρήνης, νέες, ε, νέοι κανόνες εμπορικοί. Τα πλεονάσματα τα εμπορικά έκτοτε, όπως ξέρετε, έχουν σαν συνέπεια ελλείμματα άλλων. Δεν μπορεί να περιοριστούμε σε αυτάρκεια. Και βεβαίως εδώ είναι και θέματα εθνικής κυριαρχίας, εθνικής ανεξαρτησίας και επιδοτήσεων, οι οποίες επιτρέπονται σε κάποιες περιπτώσεις. Απαγορεύεται όμως το ντάμπινγκ και είναι σαφές ότι σήμερα η Κίνα δεν είναι μια οικονομία της αγοράς, είναι μια οικονομία που προστατεύεται και βεβαίως δεν ασχολείται με τα συμφέροντα των άλλων χωρών. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ίσες εμπορικές συναλλαγές με την Κίνα και να επανέλθουμε στις θεμελιώδεις αρχές του χάρτη της Αβάνας. Πρόκειται για θέματα διεθνούς εμπορικής ισορροπίας μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βρούμε λοιπόν βιώσιμες εμπορικές συναλλαγές και αυτό θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια του ΟΗΕ και όχι του ΠΟΕ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και τώρα για ένα 1,5 λεπτό ο Σιλβαντορετσίκου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι όλοι συμμεριζόμαστε το γεγονός ότι η Κίνα, παρά το γεγονός ότι έκανε μεγάλη πρόοδο ως προς τις υποχρεώσεις της, είναι ελληματική και υπάρχουν θέματα σοβαρά που εκκρεμούν. Πιστεύω ότι οι ξένες επιχειρήσεις δεν μπορούν να δράσουν. Υπάρχει προστατευτισμός από την κυβέρνηση και κυβερνητικός παρεμβατισμός. Άρα το ερώτημά μας είναι ζωτική σημασία. Μπορούμε να χορηγήσουμε το καθεστώς οικονομίας της αγοράς στην Κίνα το Δεκέμβριο του 2016. Εάν γίνει αυτή η αναγνώριση, τότε η Κίνα θα προκαλέσει μια μεγάλη έλλειψη θέσεων εργασίας στο δικό μας βιομηχανικό τομέα. Δεν θα υπάρχει προστασία της εργασίας, θα υπάρχει μείωση εργασίας κατά 30-50%. Θα θέλαμε λοιπόν να υπάρχουν εγγυήσει για να μπορέσουμε να χορηγήσουμε αυτό το καθεστώς και θα θέλαμε να ξέρουμε τη στρατηγική της Κομισιόν έτσι ώστε να εξασφαλίσει και να διασώσει θέσεις εργασίας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτοματισμούς, ούτε μερικές επαληθεύσεις των επιπτώσεων αυτής της αναγνώρισης. Σήμερα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πικρή αλήθεια. Τι μπορεί να συμβεί. Χρειάζεται ένα αριθμιστικό πλαίσιο, αλλά θα θέλαμε αυτή τη στιγμή να υπάρξει μία ρυθμιστική και υπεύθυνη θέση. Ο Βίκτορ Μποστινάρου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι ένα πολύ λεπτό θέμα και είναι σημαντικό να καταλάβουμε την ουσία του καθώς και τις συνέπειες και της μίας και της άλλης επιλογής η συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής είναι απαραίτητη και ουσιώδης. Βλέπουμε ότι από οικονομικής απόψεως οι εμπορικές αυτές συναλλαγές είναι πάρα πολύ σημαντικές και για τα δύο μέρη. Το ίδιο όμως σημαντικό είναι και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και βιομηχανίας. Και αναφέρθηκα στην συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής, γιατί βεβαίως η εμπειρογνωμοσύνη, οι έρευνες, οι μελέτες αντικτύπου της Επιτροπής είναι αυτές που μπορεί να οδηγήσουν στην σωστή απόφαση. Και εδώ σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να δημιουργηθεί αντιπαράθεση ή εμπορικός πόλεμος μεταξύ ημών και της Κίνας. Όλα τα μέτρα θα πρέπει να εξεταστούν έτσι ώστε να αποφύγουμε ένταση και επιπτώσεις αρνητικές για την οικονομία μας, τις επιχειρήσεις μας και την απασχόληση. Νέα εργαλεία. Σας ευχαριστώ πολύ, ο Μπάς Μπέλτερ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η αναγνώριση του καθεστώτος οικονομίας της αγοράς στην Κίνα έχει μεγάλη συνέπειες όπως ακούσαμε και στη Χαλιδευουρία και αλλού διακυβεύονται πάρα πολλές θέσεις εργασίας και δεν γίνεται λόγος για αυτόματη αναγνώριση. Καλά θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να δει τι γίνεται με τον Καναδά και την Αυστραλία και πώς ε, δόθηκε ε, το καθεστώς στις χώρες αυτές ε, σταδιακά, βαθμιαία σε συγκεκριμένους κλάδους της βιομηχανίας που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις. Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Επίσης, θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση ε, των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην Κίνα, να δούμε τι γίνεται με τις ε, εξαγωγές. Παρακαλώ να μην απογοητεύσετε, κυρία Επίτροπε, τις δικές μας επιχειρήσεις και τους εργαζομένους. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό επίσης, η Ντίτα Χαράντσοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η δυνατότητα χορήγησης του καθεστώτος οικονομίας της αγοράς στην Κίνα αναφέρεται όλο ένα και περισσότερο. Ακόμα και σε μας την τσεχική δημοκρατία, όπως είπατε, δεν έχει μόνο νομική υπόσταση αυτό το θέμα. Θα έχει και οικονομικές επιπτώσεις και χαίρομαι που προσδίδεται την δέουσα σημασία σε αυτό το ζήτημα. Αναφερθήκατε ε, σε υποθέσεις προηγούμενης εβδομάδας που θα αναφέρεται και στο ε, Συμβούλιο Υπουργών Εμπορίου. Αλλά θα πρέπει να έχουμε μία ε, καλύτερη μελέτη επιπτώσεων. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο Β. Τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση εάν η Κίνα αποκτήσει το καθεστώς οικονομίας της αγοράς και ποια μέσα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να προστατεύσουμε το μης από ανταγωνισμό. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα πρέπει να δοθεί το καθεστώς της uh, οικονομίας αγοράς στην Κίνα αυτή τη uh, στιγμή. Καθότι δεν καθορίζονται ελεύθερα από την αγορά ούτε οι τιμής, ούτε υπάρχει κάτι το οποίο δεν ελέγχεται και δεν επιβάλλεται από το πενταετές ε, κρατικό πρόγραμμα. Είδατε εξάλλου ποια είναι οι πάρα πολύ αρνητικές επιπτώσεις ε, στον τομέα του Χάλιβα για το Ηνωμένο Βασίλειο και για άλλες χώρες της πολιτικής και των εξαγωγών της Κίνας. Βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται κάτι τέτοιο και ότι κάθε φορά που υπάρχουν επιδοτούμενοι τομείς καθώς και το ε, πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εκπομπές, κάθε φορά η πολιτική της Κίνας έχει επιβλεβεί συνέπειες για εμάς. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν πρέπει να δοθεί το καθεστώς οικονομίας αγοράς στην Κίνα. Ο κύριος Πρόντουστ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτρεπε, πρόκειται για κάτι που μας προβληματίζει και οφείλεται ουσιαστικά στη μέθοδο υπολογισμού μας. Και εδώ ουσιαστικά δεν πρόκειται για την ερμηνεία μιας φράσης, μιας διατύπωσης σε ένα νομικό κείμενο ή σε ένα ε, πρωτόκολλο. Πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο θα πρέπει να ερμηνευθεί ορθά και όχι με ασάφεια. Η Κίνα είναι μια χώρα φίλος και όταν της ε, προσάπτουμε ότι δεν αναγνωρίζει το καθεστώς οικονομίας αγοράς, απαντά με έναν τρόπο ο οποίος είναι ακόμα πιο προστατευτικός, πιο επιθετικός για μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμπεριφερθούμε με αυτόν τον τρόπο στην Κίνα. Είδατε τι έγινε με το θέμα των φωτοβολταϊκών. Είδατε ότι η Κίνα κατάφερε να διχάσει την πρώτη εμπορική δύναμη του πλανήτη μας, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε αλληλεγγύη, θα πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι, θα πρέπει να αποφύγουμε διχασμό και σε κάθε περίπτωση να δείξουμε πρώτα αλληλεγγύη προς τις επιχειρήσεις μας οι οποίες θα πληγούν από ενδεχόμενα μέτρα από μέρους της Κίνας. Θα πρέπει να βρούμε μια κοινή μέθοδο αντίδρασης και σε καμία περίπτωση να μην αντιδρούμε απλοϊκά. Δεν σας λέω ότι δεν πρέπει να αρνηθούμε κάποια πράγματα στην Κίνα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε μια αντίδραση η οποία δεν θα πλήξει τις επιχειρήσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώ Λάινεν για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Μεταξύ του να μην κάνουμε τίποτα και να έχουμε μια αυτόματη αντίδραση, ίσως υπάρχει και ένας τρίτος λόγος, μια λύση που θα ε, μας οδηγήσει σε μια πιο σωστή αντιμετώπιση της Κίνας για κάποιους τομείς και δεν θα αναφερθώ μόνο στον ε, Χάλιβα. Υπάρχουν πάρα πολλοί αρνητικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις μας από αυτές τις πρακτικές. Dumping, το dumping δεν είναι κάτι που δεν έχει συνέπειες. Είδατε ότι από την Κίνα αυτή η πρακτική μπορεί να επιδεινωθεί, να αυξηθεί. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάποια εργαλεία για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε έναντι αυτών των αθέμητων πρακτικών. Οι κινέζικες τιμές, όπως ξέρετε, είναι αδιαφανείς. Και εμείς θα πρέπει πραγματικά να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ίσο τρόπο και βάσει των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προστατευτεί... και να χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία για να το κάνει. Ευχαριστώ. οι πολυπληθείς δράσεις δείχνουν ότι η Κίνα δεν είναι πλήρως μέλος της παγκόσμιας αγοράς. Άρα δεν μπορούμε να τη μεταχειριστούμε ως τέτοια μέχρι ότου πληρεί τα πέντε κριτήρια που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να βρούμε ένα μέσο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του τομέα της χαλιβουργίας και άλλων. Και επειδή υπάρχει κρατικός παρεμβατισμός, η Κίνα προσπαθεί να ε, υπερέχει και σε άλλους τομείς. Θεωρώ ότι δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις εμπορικές ε, στρεβλώσεις αν δεν δράσουμε επαρκώς. Θα υπήρχαν ε, ολέθριες συνέπειες κατά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Εάν δεν υπάρχει μία εύρωστη πρόταση από την Επιτροπή, γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μία μελέτη αντικτύπου για να δούμε πώς μπορούμε να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα για να υπάρχουν ίσοι κανόνες πρόσβαση στην αγορά και από την Κίνα και από την Ευρώπη. Έχετε ε, μία μπλε κάρτα από τον κύριο Μίκε. Θέλετε να απαντήσετε. δέχεστε. Κόρβεν Μίκε, δέχεστε να, την να απαντήσετε. Θα ήθελα να σας πω ότι αν μπορώ να αγοράσω ένα κινέζικο αυτοκίνητο που στοιχίζει 20.000 αντί 40.000, αυτό σημαίνει ότι μπορώ να διαθέσω τα άλλα 20.000 εκεί που θέλω. Έτσι δεν είναι. Άρα τι θα γίνει με αυτό το περίσευμα. Θα πρέπει να αγοράσουν ε, αγαθά από εμάς. Δηλαδή, αν πουλήσουμε σε αυτούς, θα αγοράσουν από εμά. Έτσι δεν είναι. Κύριε Κόρβιν Μίκε, είχατε μιλήσει στη συζήτησή σας, έδωσα το λόγο έτσι καλλιώς για την ε, μπλε κάρτα, δεν κάνατε ερώτηση, κάνατε δεύτερη τοποθέτηση. Αυτά τα πράγματα δεν τα δέχομαι. Κύριε, ο κύριος Βαλένσα θα έχει την ευκαιρία να δράσει τα όσα είπατε. Thank you. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακριβώς αυτό θα έλεγα και εγώ, ότι δεν ήταν ε, ερώτηση προς εμένα αυτή. Και ο συνάδελφος δεν έχει επικοδομητικές απόψεις, θέλει να καταβαραθρώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό δεν βλέπω το λόγο γιατί να το απαντήσω. Και τώρα για ένα λεπτό η κυρία Μαρία Γενά. Ευχαριστώ. Όπως είπαν και οι συνάδελφοί μου, είμαστε κατά της αυτόματης χορήγησης ε, του καθεστώτος οικονομίας αγοράς στην Κίνα, θα δει ότι δεν είναι οικονομία της αγοράς και θα πρέπει να το λέμε. Ακόμα και αν ορισμένοι φρονούν ότι δεν είναι αυτό το θέμα, όχι, η Κίνα δεν είναι οικονομία αγοράς. Από την άλλη θέλουμε αποτελεσματικά εργαλεία κατά του ντάμπινγκ απέναντι στον αθέμητο ανταγωνισμό και θέλουμε να διατρανώσουμε επίσης ότι η λύση που θα πρέπει να βρεθεί δεν θα πρέπει να είναι τομεακή, γιατί γίνεται μεγάλος λόγος για τη χαλιβουργία, αλλά δεν είναι ο μόνος τομέας, ο μόνος κλάδος που σήμερα θίγεται και πλήττεται από αυτή την επιθετική στάση της Κίνας. Ε, ούτε θέλουμε κάτι που να συνδέεται με ειδικά συμφέροντα κάποιων κρατών μελών. Ε, θέλουμε αποτελεσματικά μέσα, όχι προστατευτισμού όπως ορισμένοι είπαν, αλλά απλούστατα προστασίας απέναντι σε επιθετικές και αθέμητες ε, πρακτικές της Κίνας σήμερα. Ευχαριστώ. Εξαιρετικός από χρόνο ο λόγος σας ο κύριος Φαντεγκάμπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ καταρχάς την Επίτροπο για την πάρα πολύ προσεκτική διαδικασία που τήρησε και την ενημέρωση που πήραμε απόψε ως μέλος της Αντιπροσωπείας για την Κίνα και ως μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, αλλά και ως Ολλανδός, ε, έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι για να υπάρξει καλή εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας θα πρέπει να καταλάβουμε ε, ότι θα πρέπει η Κίνα να αναπτυχθεί και να γίνει μια γνήσια οικονομία της αγοράς. Έχουμε συμφωνίες του ΠΟΕ, έχουμε πέντε κριτήρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση συμπληρωματικά, αλλά εάν η Κίνα δεν παίζει το παιχνίδι, εμείς τι να κάνουμε. Εμείς ε, δεν μπορούμε να απαιτούμε από τους ψηφοφόρους και τους λαούς μας ε, να υφίσταται και ε, το ντάμπινγκ των φωτοβολταϊκών και της χαλιβουργίας. Εύχομαι στην Επίτροπο καλή τύχη, στην προσεκτική ε, μελέτη αντικτύπου. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, αλλά διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Ευχαριστώ για ένα λεπτό, Γιάχιμ Σούστερ. Κύριε Πρόεδρε, το ελεύθερο εμπόριο έχει ε, όφελος μόνο όταν είναι δεδομένοι οι ε, κανόνες του παιχνιδιού και ο δίκαιος ανταγωνισμός και ο θεμητός. Αυτό δεν το κάνει η Κίνα. Αυτό το βλέπουμε ε, στις αγωγές χαλιβουργίας στην Ευρώπη. Ε, έχουμε πολλές ε, επιχειρήσεις που εδρεύουν εδώ και κινδυνεύουν ε, μαζικά και απειλούνται θέσεις απασχόλησης. Αν δοθεί το καθεστώς ελεύθερης οικονομίας στην Κίνα θα είναι πολύ πιο δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τέτοιες πρακτικές. Είναι προφανές ότι η Κίνα δεν είναι οικονομική οικονομία της αγοράς. Αλίμονο. Και υπάρχουν και πολύ λίγα σημάδια ε, ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να εγκαταλείψει ε, ή να αλλάξει τις κρατικές επιχορηγήσεις και τη σχεδιαζόμενη οικονομία. Όλα ε, συγκλίνουν προς την κατεύθυνση ότι θα συνεχιστεί αυτό. Το θέμα δεν είναι προστατευτισμός νέου, είναι οι δίκαιοι κανόνες του εμπορίου και εκεί καλείται και η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξηγήσει πώς θέλει να αντιδράσει στο ντάμπινγκ. Και κυρία Επιτροπέ πρέπει να σας πω ότι με έχετε απογοητεύσει λίγο. Σήμερα δεν είπατε τίποτα συγκεκριμένο τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα λεπτό τώρα, Φιέλνερ. Ευχαριστώ πολύ. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι για πολλούς είναι ένα ιδεώδες η οικονομία της αγοράς. Το επιχείρημα όμως αυτό δεν αρκεί. Το θέμα δεν είναι αν είναι ή δεν είναι η Κίνα η οικονομία της αγοράς. Το θέμα είναι αν εμείς θέλουμε να τηρήσουμε και να σεβαστούμε το ότι η Κίνα είναι μέλος ε, του ΠΟΕ και αν θέλει ως μέλος του ΠΟΕ να σεβαστεί και να τηρήσει τους κανόνες που διέπουν τον οργανισμό αυτό. Βεβαίως υπάρχουν συνέπειες για την απασχόληση. Δεν το έθιξε όμως αυτό η Επίτροπος και βεβαίως ε, η αναθεώρηση των μέτρων κατά του ντάμπινγκ ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι που μας απασχολεί. Εδώ χρειαζόμαστε μια πρόταση που να σέβεται τους κανόνες, που να μην βάζει επιπλέον εμπόδια για την Κίνα και βεβαίως να δημιουργεί μια προστασία κατά του ντάμπινγκ. Καλή τύχη! Ευχαριστώ πολύ. Ο Εμμανουέλ Μορέλ για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως έλεγε ο Ντέβιντ Μάρτιν, υπάρχει θέμα πρόβλεψης. Επί 15 χρόνια ξέρουμε ότι το θέμα αυτό μπορεί να προκύψει και τώρα μέσα σε πανικό προσπαθούμε να βρούμε μέσα για να αντιμετωπίσουμε κάτι που ξέραμε θα έρθει. Η Κίνα δεν είναι η οικονομία της αγοράς. Εξάλλου, όταν κάποιος μιλάει με Κινέζους, δεν θεωρούν ότι υπάρχει οικονομία αγοράς στην χώρα τους. Το θέμα λοιπόν είναι δικό μας. Εμείς τι Ευρώπη επιθυμούμε. Μια Ευρώπη η οποία έχει ιδέες, η οποία οραματίζεται πράγματα, μια Ευρώπη που προστατεύεται. Έχω την εντύπωση ότι σε καμία περίπτωση δεν ισχύει αυτό που λένε κάποιοι συνάδελφοι, ότι αν εμείς βοηθήσουμε την Κίνα θα μεταρρυθμιστεί πιο γρήγορα. Αυτό δεν ισχύει και ας μην είμαστε ο αφελής. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προστατευτούμε, γιατί είναι σίγουρο, κυρία Επίτροπε, νομίζω καταλάβατε τι λέμε, δεν υπάρχει περίπτωση να δώσουμε το καθεστώς σήμερα στην Κίνα της οικονομίας αγοράς. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό. Έχει το λόγο κυρία Κρίτον Ντάρλινγκ. Ξέρουμε ότι αυτή η απόφαση θα έπρεπε να ληφθεί κάποια στιγμή. Το περιμέναμε εδώ και 15 χρόνια όταν μπήκε η Κίνα στον ΠΟΕ. Αλλά κανένας εδώ δεν είπε ότι η Κίνα είναι η οικονομία της αγοράς. Η δική μου ε, εκλογή, στη δική μου εκλογική περιφέρεια γνωρίζουν τι γίνεται με το dumping, πώς έχει πληγεί η χαλιβουργία μας. Το ξέρει αυτό ο μέσος ψηφοφόρος της επικράτειάς μου. Περιμέναμε εδώ και χρόνια να γίνει ένας εξυγχρονισμός. Εμείς προβάλλουμε μία ε, μειοψηφία, μία αναστέλουσα μειοψηφία στο Συμβούλιο και φαίνεται ότι εσείς χύνετε κροκοδίλια δάκρυα, κάνετε συμφωνίες με την Κίνα, αλλά δεν προωθείτε μία πρακτική ε, αντιμετώπισης και προστασίας για τη δική μας χαλιβουργία. Έχετε μία μπλε κάρτα, την δέχεστε. Ευχαριστώ. Μπορεί η συνάδελφος να δέχτε ότι στη βορειοανατολική Αγγλία υπάρχουν εξαγωγές προς την Κίνα πολύ περισσότερες από άλλες ε, περιοχές της Αγγλίας. Και επίσης ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ξέρετε ότι το εμπόριο του σκραπ έχει, βρίσκεται στα χέρια πέντε επιχειρήσεων, αν λάβουμε υπόψη και τον αποδεκατισμό της Χαλιβουργίας. Ευχαριστώ, Τζόναθαν, για την ερώτησή σου. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέρος ε, της λύσης για το τομέα της ε, Χαλιβουργίας και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ένα συνολικό σχέδιο για την ανακύκλωση ε, του, του σκράπ Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει το θέμα αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Πολλά μπορούμε λοιπόν να κάνουμε και θα πρέπει να προωθήσουμε και το εμποριό μας και τη δική μας χαλιβουργία. Η κυρία Χάντς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι η Κίνα δεν μπορεί παρά να πάρει αυτό το καθεστώς της οικονομίας αγοράς. Καλύπτει ε, ένα από τα κριτήρια που έχουμε θέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως υπάρχει και το πρόβλημα όλων αυτών των τομέων που πλήττονται από τις εξαγωγές της Κίνας και για τις οποίες είναι, απαραίτητες να είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα κατά του ντάμπινγκ. Και αυτό με όλα τα μέσα. Αναφέρομαι ιδιαίτερα και στον τομέα του χάλιβα, του γυαλιού, των κεραμικών και πολλούς άλλους τομείς που πλήττονται από τα προϊόντα της Κίνας και της Κινέζικης τιμές. Θέλουμε μια ίση μεταχείριση και αν θέλει η Κίνα πραγματικά να πάρει το καθεστώς της οικονομίας αγοράς θα πρέπει να λειτουργήσει με ένα σύγχρονο τρόπο και σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταία ομιλήτρια στην κανονική συζήτηση. Για ένα λεπτό το λόγο έχει η Ματκουλάδα Ροτρίγκε Πινιάρου Φερνάνδη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε, η πραγματικότητα είναι διαφυσβήτητη. Το Δεκέμβριο του 2016 γνωρίζουμε ότι η Κίνα δεν πρόκειται να είναι η οικονομία τη αγορά, και ειλικρινά δεν νομίζω ότι θα σταματήσει ούτε να επιδοτεί την παραγωγή, ούτε τι τιμέ, ούτε να κάνει ντάμπικ, ούτε τίποτα, ούτε το κράτο θα σταματήσει να ανακατεύεται στην οικονομία. Είναι γεγονό ότι είναι μεγάλη εμβέλεια η πολιτική απόφαση. Όλοι υφιστάμεθα πιέσει των εκπροσώπων των κινέζικων θεσμών. Αλλά ε, η πίεση δεν σημαίνει ότι έχουν και δίκιο. Η εμπορική πολιτική δεν θα πρέπει να είναι εχθρός της βιομηχανίας μας. Καινοτόμοι τομείς ε, απειλούνται γιατί η Κίνα δεν τηρεί τους κανόνε και κάνει dumping. Και γιατί μπορεί αυτό να απειλεί σοβαρά ε, εκατομμύρια ολόκληρα οικογενειών και θέσεων εργασίας. Και δεν μιλώ μόνο για τις άμεσες και για τις έμεσες θέσεις εργασίας. Η χαλιβουργία, η κεραμική που στην περιοχή μου απασχολεί πάνω από 27.000, απειλείται. Θα πρέπει να γίνει αυτή η μελέτη αντικτύπου που όλοι ζητήσαμε και σας παρακαλώ μια συντονισμένη πολιτική με τους εταίρους μας έτσι ώστε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην λάβει απόφαση μόνο μέρη. Ευχαριστώ. Και τώρα ερχόμαστε στη διακρισία Κατσέη. Η κυρία Σόιντροβα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε, συνάδελφοι, νομίζω ότι ακούσαμε την υποστήριξη της Επιτροπής σε σχέση με την προπαρασκευαστική εργασία για το επόμενο έτος για να προστατεύσει την ευρωπαϊκή αγορά από το κινέζικο ντάμπινγκ. Όμως άκουσα με μεγάλη έκπληξη την Επιτροπή να λέει ότι η Κίνα δεν είναι η οικονομία της αγοράς. Αυτό αντιτίθεται με ότι προελέχθη από μερικούς εδώ. Αναφέρθηκε ότι δεν μπορούμε παρά να την Κίνα ως οικονομία της αγοράς διότι έχει λήξει η 15 ετής περίοδος. Τι νόημα έχει αυτή η 15 η περίοδος εάν δεν ε, ανελήφθη η δραστηριότητα. Να προστατέψουμε την ευρωπαϊκή αγορά και βλέπουμε όλοι ότι υπάρχει κίνδυνος και κοινωνικού ντάμπινγκ και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και άλλα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να ανατρέψουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ. Εσάς Κουμπιλπάου, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η Κίνα δεν είναι η οικονομία της αγοράς, ε, ούτε στις ε, διάφορες συνθήκες εργασίας, οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές, όλα αυτά δεν είναι συμβατά με αυτά που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά ευνοούν το ντάμπινγκ και τώρα στη χώρα των Βάσκων και σε άλλες περιφέρειες ε, απειλείται η χαλιβουργία και η ε, χαλιβουργία και τα συνεφή επαγγέλματα κινδυνεύουν. Το μέλλον τους απειλείται. Οι θεσμοί μας ε, είναι ε, σε συναγερμό. Η Ευρώπη δεν θα πρέπει να καταστρέψει αυτή τη βιομηχανία. Η Κίνα χρειάζεται μεταρρυθμίσεις και θα πρέπει να γίνουν αυτές σε βάθος. Χρειαζόμαστε ε, αναδιανομή πλούτου, παγκοσμίω, κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη είναι τοξική η κατάσταση εργασιακή που επικρατεί στην Κίνα, αυτά τα μεσονικά πράγματα, όσο τοξικό είναι και το νέφος που καταγγέλουμε καθημερινά στο Πεκίνο. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Συνεχίζει ο κύριος Καπούτο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Αυτή είναι η πρώτη μας ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε το θέμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε μελέτη αντικτύπου για να δούμε τα ενδεχόμενα σενάρια, τομεακά και γεωγραφικά, έτσι ώστε να προβάλλουμε μια στρατηγική αντι-dumping. Θα πρέπει η Επιτροπή να προβεί σε δημόσια διαβούλευση με βάση νομοθετικές πρωτοβουλίες για να συνεισφέρουμε όλοι επειδή αύριο το Συμβούλιο Υπουργών Εμπορίου θα ασχοληθεί, θα πρέπει να μιλήσουμε για 210.000 θέσεις εργασίας που θα καταργηθούν. Αυτά λένε οι εκτιμήσεις. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να χορηγηθεί το καθεστώς αυτό στην Κίνα μόνο εάν πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και να υπάρχει και ένα σχέδιο Β για να υπάρχουν ε, ισοδύναμα μέτρα εάν χρειαστεί. Ο κύριος Μαριάς για ένα λεπτό. Η συζήτηση σχετικά με το καθεστώ τη κινεζική οικονομία συνδέεται άμεσα με το κατά πόσο θα μπορούν να συνεχίσουν να επιβάλλονται σε βάρος των κινέζικων προϊόντων δασμοί αντι-dumping για την προστασία τη Ευρωπαϊκή χαλιβουργίας και άλλων βιομηχανιών. Όμω πριν να συζητηθεί αν υπάρχει ή όχι η οικονομία τη αγορά στην Κίνα θα πρέπει να συζητηθεί η σταδιακή κινεζοποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας αφού καιρό τώρα οι ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρούν να μιμηθούν τις αντίστοιχες κινεζικές στα ζητήματα διαχείρισης και εργασιακών δικαιωμάτων. απόδειξη της ουσιαστικής σύγκλησης συμφερόντων η ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης του οργανισμού λιμένος Πυραιός, που προωθεί το ταϊπέδ με το ξεπούλημα της τελευταίας προβλήτας που παρέμεινε σε δημόσιο έλεγχο άνευ διαμαρτυριών από πλευράς τρόικας και δανειστών η δίθεν αυτή επένδυση στους κινέζους προσφέρει, που προσφέρουν 368 εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο όταν τον περασμένο χρόνο αγορά αντίστοιχου τουρκικού θερματικού ίδιας δυναμικότητας από την ίδια κινεζική εταιρεία κόστισε 800 εκατομμύρια ευρώ. ευχαριστώ. Ο Τάκουλα για λεπτό. Ευχαριστώ. Όπως ακούσαμε σε αυτή τη συζήτηση, η Κίνα δεν είναι η οικονομία της αγοράς. Και βεβαίως συζητάμε αν ναι ή όχι πρέπει να τους δώσουμε αυτό το καθεστώς. Νομίζω όχι. Και αυτό διότι καταρχήν πρέπει να στηρίξουμε τη χώρα αυτή προς τον εκδημοκρατισμό, προς το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προς την προστασία του περιβάλλοντος, όμως το dumping, ιδιαίτερα στον τομέα του χάλιβα, είναι κάτι που μας ε, δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι η Κίνα θα αρχίσει επιτέλους να σέβεται κοινέ αξίες και να λειτουργεί με αρχές της δεν θέλουμε πλήρη ελευθερία στην αγορά τους. Όμως να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, τους οποίους να σέβεται η Κίνα. Μπορούμε να βοηθήσουμε λοιπόν την Κίνα να πάει προς αυτή την κατεύθυνση έτσι ώστε κάποια στιγμή να τους δοθεί αυτό το καθεστώς της ελεύθερης οικονομίας. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Πρόεδρε. Majority Βεβαίως, στην ε, δική μου επικράτηρα, στην ε, Ουαλία, το θέμα αυτό μας απασχολεί. Η δική μου πολιτική δύναμη, το κόμμα μου, θέλει και προσπαθεί να σώσει το τομέα του χάλιβα στην Ουαλία. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπάρξει μια πραγματική έρευνα του τι γίνεται στην Κίνα και όχι μια εντάχει ε, μελέτη, μια κοινή και μεθοδευμένη αντίδραση μας χρειάζεται. Διότι σήμερα βλέπουμε ότι απειλούνται στην ε, Ουαλία χιλιάδες ε, ακόμα θέσεις απασχόλησης. Το καθεστώς της οικονομίας αγοράς καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερες δυσκολίες. Δεν θα μπορέσουμε να επιβάλλουμε απολύτως κανένα περιορισμό στις εξαγωγές της Κίνας. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταία μιλήτρια, κυρία Μπέγκιν. Grazie, Κυρία Επίτροπε, εμείς στο παρελθόν είχαμε ζητήσει από την Επιτροπή μία τεχνική μελέτη σε σχέση με τη χορήγηση του καθεστώτος ε, οικονομίας της αγοράς στην Κίνα. Δεν περίμενα να πολιτικοποιηθεί το θέμα. Μιλάτε για 230.000 θέσεις που θα καθούν. Εμείς μιλάμε για 3 εκατομμύρια. Αυτά λένε οι ανεξάρτητες μελέτες. Γιατί υπάρχει τέτοια διαφορά. Εσείς λέτε ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε γιατί μόνο 1,38% των ε, εξαγών από την Κίνα υφίστανται δασμούς. Μα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όταν ο δασμός πια, όταν οι δασμοί δεν θα ισχύσουν, τι θα συμβεί. Γιατί να μην κάνουμε έναν υπολογισμό πριν από τα μέτρα αντι-dumping. Επίσης, δεν μιλήσατε παρά για την χορήγηση του καθεστώτος. Δεν μιλήσατε για δασμούς αντι-dumping. Νομίζω ότι από αυτή τη μελέτη είναι σαφής οι προθέσεις της Επιτροπής που δεν, που δεν είναι καθόλου καλές για τους εργαζόμενους. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε τη διαδικασία Catch Η κυρία Μάλστρομ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους. Άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά τα μηνύματα που στέλνετε προς την Επιτροπή. Φυσικά και γνωρίζει η Επιτροπή το πόσο περίπλοκο είναι το θέμα αυτό και βεβαίως τις επιπτώσεις για κάποιους τομείς και για τις θέσεις απασχόλησης. Αυτό που κάνουμε σήμερα βεβαίως είναι να αντιμετωπίζουμε τις παρούσες τρευλώσεις της οικονομίας και βλέπουμε ότι η Κίνα αυξάνει την παραγωγή, δημιουργώντας ακόμα περισσότερες δυσκολίες. Και βεβαίως ε, η Επίτροπη, οι συνάδελφοί μου και εγώ θέλουμε να έχουμε επαφές με την Κίνα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συνεχίζουν να πλημμυρίζουν τις αγορές μας με φτηνό χάλιβα. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο το πώς θα εξελιχθούν αυτές οι συζητήσεις, για το αν ναι ή όχι θα δοθεί το καθεστώς της οικονομίας αγοράς. Υπάρχουν πολλές λοιπόν πτυχές και είναι περίπλοκο το θέμα. Υπάρχουν και οι νομικοί οι οποίοι εργάζονται για να καλύψουν τους υπόλοιπους τομείς και για να συνεχιστεί η εισβάθος μελέτη του θέματος αυτός. Πρόκειται για εκατομμύρια βεβαίως θέσεις απασχόλησης και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το καθεστώς. Έτσι κι αλλιώς και άλλοι τομείς πλήττονται και εδώ αναφερόμαστε στο 1,35% των εμπορικών μας συναλλαγών με την Κίνα που πλήττονται από αυτό το dumping. Δεν είναι όλες οι υπόλοιπες συναλλαγές. Οι αθέμητες λοιπόν πρακτικές οι οποίες ε, προέρχονται από την Κίνα βεβαίως απειλούν ε, θέση απασχόληση στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλουμε να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με την Κίνα, να τηρούνται κοινοί κανόνες και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα επόμενο θέμα αυτό.